I Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Και παρόλο που είμαι βουλευτής από το Ενωμένο Βασίλειο, η γερμανική μου παράδοση και κουλτούρα μου επιτρέπει να επιμένω στην συνέπεια στην ώρα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να καλωσορίσω τον Γέρζη Πομιανόφσκι. Ελπίζω να το πρόφερα σχετικά σωστά. Σημείο 7 στην ημερήσια διάταξη, ανταλλαγή απόψεων με τον Γέρζη που είναι εκτελεστικός διευθυντής της, του Ευρωπαϊκού Καταπιστεύματος για τη Δημοκρατία. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην Επιτροπή μας Γέρζη. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας σήμερα για να δούμε τα θέματα που απασχολούν ε, τη δημοκρατία σε μια στιγμή που δέχεται πολλές πιέσεις η δημοκρατία σε όλο τον κόσμο. Έχουμε μια κοινή πρωτοβουλία λοιπόν που ξεκίνησε από το 2013 με το καταπιστευμό από, την, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Η πρώτη απόφαση λήφθη το 2011 και έκτοτε υπήρξαν πολλές εξελίξεις, αλλαγές και ε, διακυμάνσεις στο διεθνές προσκήνιο. Πιο συγκεκριμένα, ο οργανισμός σας στηρίζει μια, ε, ένα ευρύ φάσμα ε, φορέων οργανώσει τη κοινωνίας των πολιτών, ακτιβιστές, ανεξάρτητες πλατφόρμες μέσων μαζικής ενημέρωσης, δημοσιογράφους που εργάζονται για ένα πολυφωνικό πολιτικό σύστημα. Εδώ συμπεριλαμβάνονται και μη εγγεγραμμένες οργανώσεις, ελεύθερες οργανώσεις, ιδιώτες και άλλου είδου σύλλογοι και ενώσει. Ε, ένα πρώτο σημαντικό πράγμα είναι η υποστήριξη αυτών που δεν μπορούν να υποστηριχθούν από άλλους δωρητές ή από άλλα εργαλεία της Ένωσης. Προσφέροντας χρηματοδότηση και που υπάρχουν δυσκολίες για οποιαδήποτε άλλη χρηματοδότηση με τις κλασικές διαδικασίες. Είναι σημαντικό για την υποεπιτροπή μας να δούμε από την αρχή της κοινοβουλευτικής μας θητείας πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σταθερή σχέση συνεργασίας και με και με, άλλους, του όλους τους οργανισμούς που ασχολούνται με τα θέματα των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε περιφερειακό και διεθνέ επίπεδο. Τα μέλη της Επιτροπής μας θα ήθελαν τις απόψεις σας για τις τάσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση Ανατολικά και Νότια, αλλά και στη Μέση Ανατολή, στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Τουρκία, και το απόψεις σας για τις διάφορες συγκρούσεις και τις μεταβατικές καταστάσεις. Ξέρουμε ότι ενεργοποιήσετε και σε άλλες χώρες όπως το Μπαχρέιν, το Τσάντ, το Ιράν, το Ιράκ, το Ισραήλ, το Κουβέιτ, το Μαλί, ε, η Νιγηρία, το Κατάρ, το Ομάν, ο Νίγηρας, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Τζαγκιστάν, το Τουρκμενιστάν και το Ουσμπεκιστάν μεταξύ άλλων. Μπορείτε να μας πείτε πώς μπορούμε να εργαστούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για, ένα για μια συντονισμένη προσέγγιση στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Κύριε Πομιανόφσκι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για την πρόσκλησή σας και για την εισαγωγή αυτή. Ευχαριστώ την υποεπιτροπή σας που αφιερώνει χρόνο στο να ακούσει τις πληροφορίες που έχει να δώσει το δικό μας καταπίστευμα. Ελπίζω ειλικρινά αυτή η πρώτη εμφάνισή μας να μην είναι και η τελευταία. Θα εξηγήσω στη συνέχεια ότι με πολύ μεγάλη ικανοποίηση ε, θέλουμε να σας βοηθούμε και ακριβώς όποτε μπορούμε να σας δίνουμε πληροφορίες, η ανάλυση μας ικανοποιεί πάρα πολύ. Ή όταν σας υποστηρίζουμε ε, Ε, βουλευτές και οργανώσεις με τις οποίες συνεργάζεστε στα πλαίσια της εντολής μας. Υπό την έννοια αυτή έχω μεγάλες προσδοκίες ε, και φιλοδοξώ να έρχομαι πιο συχνά ή να σας δώσω την ευκαιρία να συναντηθείτε με ορισμένα μέλη της ομάδας μου, συνεργάτες που ειδικεύονται σε συγκεκριμένες χώρες και περιφέρειες για να έχετε πιο λεπτομερή πληροφόρηση. Σήμερα θα προσπαθήσω να σας δώσω μια γενικότερη εικόνα ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι νέα κοινοβουλευτική περίοδος και μπορεί ορισμένοι από εσά να μην γνωρίζουν τα, τις δράσεις μας και τη, της λειτουργίας και της ε, σύνθεσης μας. Εχθές είχα την ευκαιρία να σας πω να συναντηθώ με την κυρία Μαρία Αρενά, την πρόεδρό σας, και της έδωσα επίσης πολλές λεπτομέρειες γνωρίζω ότι σήμερα έχει άλλες ανελημμένες υποχρεώσεις. Ταυτόχρονα το καταπίστευμά μας συνεχίζει να έχει διάλογο με ένα σημαντικό τμήμα ε, του συστήματος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδιαίτερα να αφαιρθώ εδώ στον ειδικό απεσταλμένο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι ο κύριος Σίμων Γκίλμορ αυτό τον καιρό και είχα την ευκαιρία να συναντηθώ μαζί του και συντονίζουμε πολύ τη δράση μας. Έχει σημασία να πούμε το εξής το καταπίστευμα για τη δημοκρατία. Δεν ε, ε, εκπροσωπεί συμφέροντα. Ε, υποστηρίζουμε διάφορους δικαιούχους και αυτός είναι ο βασικός μας ρόλος και δουλειά μας. Καμιά φορά μπορεί να μην φαινόμαστε στη δράση μας, γιατί κυκλοφορούμε κάτω από τα ραντάρ, ούτε από την ιστοσελίδα μας, ούτε από σημαντικές δηλώσεις μπορείτε να βρείτε τι κάνουμε. Γι' αυτό προσβλέπουμε πάρα πολύ στη δική σας Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προβολή μας. Ε, όλοι εκείνοι που έχετε πολιτική φωνή και ακούγεται ε, να θέτετε αυτά τα ζητήματα. Ε, πάντως, κάθε φορά που συναντιόμαστε και αν θέλετε ε, την ειδική υποστήριξη που μπορούμε να σας δώσουμε, αυτό μπορεί να γίνει σε πιο διμερή μορφή όταν συζητούμε για ευαίσθητα έργα. Από την αρχή, όπως ακούσαμε προηγουμένως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ακρεφνής υποστηρικτής του καταπιστεύματός μας και ήταν και από τα θεσμικά όργανα που πίεζαν για την ίδρυσή μας το 2012 και 2013, όταν άρχισε να λειτουργεί η οργάνωσή μας όπως είπατε, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε ληφθεί το 2011. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως συζητούσε το ενδεχόμενο θέσπισης ενός τέτοιου ταμείου ε, θεσμού ε, από το 2006 ήδη. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση και πολύ ενδιαφέρον ε, δείχνει το Κοινοβούλιο. δεν χρειάζεται να σας πω ότι εννέα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του καταστατικού μας είναι μέλη και του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Κάθε φορά λοιπόν που εκλέγεται ένα νέο κοινοβούλιο ε, ορίζει εννέα, ε, εννέα μελή αντιπροσωπεία ε, που αναλαμβάνει μέλος στο δικό μας Διοικητικό Συμβούλιο. Εκεί έχουμε εκπροσώπους των κρατών μελών που συνεισφέρουν και συμμετέχουν στο καταπίστευμα έχουμε εκπροσώπους από άλλους θεσμούς, την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε και μια τριμελή εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Πολιτών που δίνουν τη δική τους ματιά και σκοπιά ε, από οργανώσεις που στηρίζουν ε, την προσπάθειά μας στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν μεικτή εκπροσώπηση και πολιτική και θεσμική και διπλωματική και αυτό μας δίνει ε, πολύ μεγάλη ευκαιρία στο Διοικητικό Συμβούλιο να έχουμε μεγάλη πολυμορφία στις προσεγγίσεις και να δίνουμε ταυτόχρονα καλές κατευθυντήριες γραμμές στη γραμματεία και στη δράση μας. Ε, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει δις ετησίως, δηλαδή είναι πολύ φορτωμένη η ατζέντα για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιστεύουμε ότι έχει το ενδιαφέρον του αυτό γιατί κατά τη διάρκεια ε, της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο συζητώνται διάφορα ε, θέματα που επηρεάζουν άμεσα τις δράσεις μας. Πού εργαζόμαστε, ποιε είναι οι τομείς που καλύπτουμε γεωγραφικώς, ακούσαμε προηγουμένως τις χώρες. Αρχίσαμε από τις χώρες της γειτονίας, Ανατολικής και Νότιας, αργότερα η εντολή μας διευρύνθηκε και αρχίσαμε και κάποια προγράμματα στην ίδια τη Ρωσία, την Τουρκία, την Κεντρική Ασία, στους γείτονες των γειτόνων μας και προς Νότον και προς Ανατολάς, των χωρών της γειτονίας δηλαδή, και στα Δυτικά Βαλκάνια. Δεν είμαστε ακόμα παγκόσμια ε, ε, δράση εντολή μας, αλλά είναι αρκετά ευρία. ταυτόχρονα το καταπίστευμα για τη δημοκρατία δεν είναι ένας μηχανισμός που έχει στόχο να αντικαθαστήσει οποιοδήποτε υφιστάμενο όργανο. Για αυτό, από την αρχή στο Διοικητικό Συμβούλιο τονίσαμε ότι θα πρέπει να έχουμε συμπληρωματικότητα, να αποφύγουμε ε, τις επικαλύψεις και να βρούμε ε, που είναι ο δικός μας ειδικό ρόλος. Όπως φαίνεται και από το όνομα, υποστηρίζουμε τη δημοκρατία. Δεν χρειάζεται ε, να πούμε πώς αυτό επικαλύπτεται με τις δικές σας δράσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι προφανές, αλλά υπάρχουν ειδικοί τομεί όπου προσφέρονται καλύτερα ειδικοί οργανισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν υποστηρίζουν τους ε, αγωνιστές και ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα μπορούσα να σας δώσω διάφορα παραδείγματα όμως για να δείτε πόσο συχνά αυτά τα δύο θεματολόγια επικαλύπτονται, συμπίπτουν ε, και σε εχθρικό περιβάλλον όταν φυλακίζονται και στερούνται τις βασικές ελευθερίες οι άνθρωποι αλλά και σε χώρες που βρίσκονται σε δημοκρατική μετάβαση όπως πολλές χώρες που ακόμα θεωρούνται δημοκρατίες. Ε, ε το γεννάστε. η ομοφιλοφιλία ή τα δικαιώματα των πολιτών δεν γίνονται σεβαστά και έχουμε τεράστιο δημοκρατικό ε, ε, έλλειμμα ή κάποιες στοιχειώδεις δημοκρατικές διαδικασίες. Ε, αυτό είναι μια σαφέστατη ένδειξη ότι το να υποστηρίζεις τους αγωνιστές της δημοκρατίας πολύ συχνά συμπίπτει με την ε, ατζέντα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό τη στενή έννοια, την παραδοσιακή χρηματοδότηση. Η χρηματοδότησή μας είναι ευέλικτη και στην αρχή ήταν πολύ ισχυρό ατού και επιχείρημα για να δημιουργηθεί ο μηχανισμός. Στην αρχή ε, ε, είχαν όλοι καταλάβει ότι τα προγράμματα υποστήριξης της δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ σημαντικά αλλά οι διαδικασίες είναι πολύ βαριές και μακροχρόνιες. Προκήρυξη, ε, ανάθεση, έγκριση, χρηματοδότηση ήταν πολύ βαριά δομή και ε, η φιλοδοξία ήταν να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός συμπληρωματικός, ε, ενώ ως προς την ταχύτητα της δράσης. Για να σας δώσω μια ιδέα, τα πιο γρήγορα έργα που εφαρμόσαμε ήταν μέσα σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης. Δεν θέλω να το παρακάνω στη διαφήμιση, αλλά η μέση ταχύτητα της ε, έκτακτης επίγουσας υποστήριξης ε, είναι δύο εβδομάδες, το πολύ τρεις. Γιατί πραγματικά είναι ταχεία η προσέγγιση μας αυτή. Βέβαια έχουμε και εμείς τους κανόνες μας και τις διαδικασίες μας που γίνονται σεβαστές γιατί έχουμε και κάποιες ανάγκες. Ε, δεύτερον, δεν έχουμε διαγωνισμούς και προκηρύξεις και ε, όταν έρχονται τα αιτήματα εμείς αντιδρούμε ιδιαίτερα όταν υπάρχουν κρίσεις. Ε, πολλοί από εσά έχετε ακούσει τις κρίσεις ότι έγινε επανάσταση στην Ισία, στην Ουκρανία και αλλού και ο κόσμος έρχεται και μας ζητάει βοήθεια και θα του είπανε ότι ο επόμενος διαγωνισμός θα προκηρυχθεί σε έξι μήνες. Μα όταν γίνονται επιτόπου διάφορα πράγματα, προς το καλό ή προς το κακό, ε, οι ανάγκες είναι επιτακτικές και άμεσες και εκεί προσπαθούμε να έχουμε την παρουσία. Ε, βέβαια δεν μπορούμε να καλύψουμε τα πάντα, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Ε, στα έξι χρόνια που λειτουργούμε, το συνολικό ποσό της υποστήριξης ήταν 60 εκατομμύρια κατά μέσο όρο. Στην αρχή ήταν λιγότερο από 10 εκατομμύρια το χρόνο, τώρα είναι ε, αρκετά πάνω από 10 εκατομμύρια. Ε, χορηγήσεις, επιδοτήσεις είναι και εδώ μιλώ μόνο για χρήματα που πηγαίνουν άμεσα στους τελικούς δικαιούχους. Για να σας εξηγήσω, εμείς δεν υποστηρίζουμε ας πούμε οργανώσεις εκδημοκρατισμού που εδρεύουν στην Ευρώπη. Δίνουμε τα χρήματα επιτόπου στους δικαιούχους στις χώρες αυτές. Εκεί που δρούνε ε, οι φορείς αυτοί είναι απόλυτη προτεραιότητα, με λίγες εξαιρέσεις όπως πάντα και αυτό σημαίνει ευελιξία να προβλέπεις και εξαιρέσεις, αλλά γενικά είναι πολύ σημαντικό αυτό ως προτεραιότητα. Αντίστοιχα, λειτουργούμε ε, στις τοπικές γλώσσες. Δηλαδή, δεχόμαστε τις αιτήσει στη γλώσσα που μιλάει ο κόσμος σε μια χώρα. Και αναλαμβάνουμε εμείς αυτό το κόστος να ε, μεταφραστούν στις γενικές γλώσσες λειτουργίας, που συνήθως είναι αγγλικά και γαλλικά. Και τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε δώσει πολύ μεγάλη προσοχή στην ουσία, στο περιεχόμενο. Κάθε βοήθεια που προσπαθούμε να δίνουμε εξαρτάται πάντα από το περιβάλλον στο πιο εχθρικό περιβάλλον τα κλασικά ε, project που υποστηρίζουμε δεν είναι τόσο προφανή. Σε χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν ας πούμε ή όπως η Αίγυπτος και πολλές άλλες που μπορεί να γνωρίζετε, μπορεί να μιλάμε και για την Ρωσία, πολλά από τα έργα μας συνδέονται άμεσα με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί ε, σε αυτές τις χώρες υπάρχουν άνθρωποι στις φυλακές και όπου το βασικά θεμελιώδη δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά και δεν προστατεύονται επαρκώς. Σε πιο δημοκρατικά περιβάλλοντα η υποστήριξή μας γίνεται πιο πολιτική. Συνδέεται περισσότερο με την ελευθεροτυπία, με ε, τον πολιτικό ακτιβισμό, ακτιβισμό πολιτικών δικαιωμάτων, ε, ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία σημαντικά. Ε, εδώ έχουμε μια τεράστια παλέτα και διαφορά στη δράση μας. Καμιά φορά αυτό οδηγεί σε σύγκριση γιατί βλέπετε τις εκθέσεις ε, και διαπιστώνετε ότι δεν έχουμε ένα ειδικό τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και υποστηρίζουμε. Είναι γεγονός αυτό. Υπάρχουν πιο ειδικοί οργανισμοί που έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο βοήθειας και πάντα ακολουθούν αυτό ε, και είναι γνωστή η προστιθέμενη αξία τους. Εμείς ε, θα πρέπει σε κάθε έργο μας, σε κάθε project να εξηγούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο τι κάναμε, γιατί και ποια είναι η υπεραξία δεν υπάρχει ε, μια εύκολη φόρμουλα, ένας μαθηματικός τύπος να εφαρμόσουμε και να αποδεικνύουμε ότι είμαστε χρήσιμοι. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα του τι κάνουμε. Τώρα εξαρτάται από τις χώρες που σας ενδιαφέρουν. Παράδειγμα, στο Λίβανο έχουμε κάποια θέματα πολιτικών δικαιωμάτων. Υποστηρίζουμε και τους σύρους πρόσφυγες, ιδιαίτερα εκείνους που δεν έχουν κανένα νομικό δικαίωμα. Και δεν μπορούν να αυτοοργανωθούν και να υποστηρίξουν τους εαυτούς τους. Ειδικά στο Λίβανο ξέρουμε ότι οι διεθνείς ΜΚΟ αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες για να λειτουργήσουν. Τους αρνούνται το νομικό καθεστώς, δεν τους αφήνουν να λειτουργήσουν. Αυτοί οι περιορισμοί λοιπόν μας κάνουν εμάς να μπαίνουμε εκεί για να δώσουμε βοήθεια. χωρίς να χρειάζεται απαραίτητος να σεβόμαστε την νομοθεσία και ε, ε, τις ρυθμίσεις των κρατών αυτών. Και αυτή είναι η προστιθέμενη αξία και το προνόμιο του καταπιστεύματος. Δηλαδή, αν αρέσει το πρόγραμμά μας στην κυβέρνηση, είμαστε και εμείς ευχαριστημένοι. Αν δεν, σημαίνει, αν δεν αρέσει την κυβέρνηση, σημαίνει ότι μας έχει ανάγκη ο κόσμος. Βεβαίως υπάρχει και η διμερή συνεργασία μέσω των πρεσβειών, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να υποκαταστήσει τη δική μας ε, λειτουργία. Γιατί οι πρεσβείες ε, που συνεργάζονται διμερώς ε, με κάποιες χώρες οφείλουν να τηρούν την νομοθεσία της χώρας. Εμείς είμαστε ΜΚΟ ε, που εδρεύουμε στο Βέλγιο. Άρα δεν ε, ε, υποκείμεθα στο διεθνές δίκαιο. Στη Βοσνία, Ερζεγοβίνη, για παράδειγμα, αρχίζουμε να υποστηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διάλογο με την νεολαία μέσω καινοτόμου θεάτρου και τέχνης. Βλέπετε, είναι πολύ ιδιαίτερες. Στο Αζερβαϊτζάν, Λευκορωσία, Τουρκία Υποστηρίζουμε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπάρχουν εδώ και χρόνια, αλλά αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στην πρόσβαση της διεθνούς χρηματοδότησης. Στην Αίγυπτο, προφανώς, υπάρχει μεγάλη διάθεση για διεθνή βοήθεια, αλλά την σταματάνε γιατί δεν θέλει καθόλου κυβέρνηση. Παράδειγμα υπάρχει το Ίδρυμα Άννα με πολιτιστικά προγράμματα και από ό,τι έμαθα πέρσι η Αιγυπτιακή κυβέρνηση ε, σταμάτησε κάθε συνεργασία. Δεν ενέκρινε κανένα πρόγραμμα στα πλαίσια του Ιδρύματος Άννα στη συνεργασία δηλαδή με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Η δική μας υποστήριξη είναι ευέλικτη και ακριβώς είμαστε κάτω από τα ραντάρ και δεν ε, δημοσιεύουμε τη δράση μας για να προστατεύουμε τους ενδιαφερόμενους και να μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους και τη δράση τους. Ποια είναι τα προβλήματα και οι προκλήσεις. Όπως σας είπα, εμείς δεν είμαστε λόμπι, δεν εξυπηρετούμε συμφέροντα ή ε, ανθρώπινα δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ποιες είναι οι τάσεις και τι λέει η κοινότητα που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Όταν θες να προστατεύεις ε, κάποιον επιτόπου δεν έχεις πάντα τα απαραίτητα ε, εργαλεία. Ε, υπάρχουν οι διμερείς συμφωνίες, αλλά οι δωρητές δεν μπορούν πάντα να δίνουν βοήθεια λόγω του πλαισίου. Μετά υπάρχει πολιτική πίεση που δεν είναι αρκετά συντονισμένη με όλη την άλλη υποστήριξη που υπάρχει. Έχουμε λοιπόν εμικτό το μήνυμα που ακούμε από τους δικαιούχους. Πώς είναι δυνατόν ο Α ή ο Β ηγέτης να παραβιάζει τόσο κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα και μετά πάει και κάνει χειραψία με τους Ευρωπαίους ηγέτες και χαριεντίζεται. Ε, ε, αυτά είναι προβλήματα ε, που μας λένε οι άνθρωποι που έχουν τις ίδιες αξίες με μας και θεωρούν ότι δεν προστατεύονται αρκετά, ότι είναι εκτεθειμένοι δηλαδή. αλλά δεν προβάλλονται αρκετά. Επίσης βλέπουμε να μειώνεται η υποστήριξη ε, και η κατανόηση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον κόσμο. Αρχίζουν συζητήσεις από τον, αρχηγό, από τον στρατηγό Αλ Σίση στην Αίγυπτο που λέει ότι τα δυτικά ανθρώπινα δικαιώματα δεν εφαρμόζονται, δεν βρίσκουν εφαρμογή στην ε, Αιγυπτιακή πραγματικότητα. Ε, και βγαίνουν διάφορα παπαγαλάκια, δημοσιογράφοι ή εμπειρογνώμονες στις τηλεοράσεις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μεταφέρουν αυτά. Αυτό το είδος αφηγήματο ε, προκαλεί διάφορες αντιδράσεις, όπως είναι αμφιβολίες, γιατί σου λέει όλος, για να το λένε αυτοί κάτι θα ξέρουν. Μήπως ισχύει και αμφισβητούνται διάφορα πράγματα που είναι ευρέως ε, διαδεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, πεπιθήσεις και αρχίζουν να αμφιβάλλουν για το γεγονός ότι είναι οικουμενικά και αδιαπραγμάτευτα τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν χωράει σχετικοποίηση, διότι ε, αν αρχίσει αυτή η αμφισβήτηση αντιτίθεται στα θεμέλια τα ίδια του σημερινού κόσμου. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν απέναντι σε αυτές εμείς δεν είμαστε think tank δεξαμενής σκέψης, ούτε κάνουμε συστάσεις για πολιτική, ούτε λόμπι είμαστε, ούτε εκθέσεις βγάζουμε, ούτε ενημερωτικά σημειώματα. Life, Απλώς έχουμε πρόσβαση στον κόσμο επιτόπου που ζει κάποιες πραγματικότητες και μας λέει τι γίνεται. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία και για σας τους Ευρωπαίους πολιτικούς και συχνά τους φέρνουμε και στις Βρυξέλλες για να γίνεται η φωνή τους ακουστή και να υπάρχει αυτή η προβολή που τους χρειάζεται τόσο πολύ. Αν μπορούσατε εσείς να τους προσφέρετε ε, χώρο και χρόνο εμείς ως καταπίστευμα με χαρά να τους φέρουμε να τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία. Αντίστοιχα, αν ταξιδέψετε στις περιοχές των χωρών αυτών όπου εμείς δρούμε, μπορούμε να σας κάνουμε ειδικά briefing, ενημερώσεις για τις καταστάσεις, για συγκεκριμένα πρόσωπα ε, που μπορεί να χρειάζεται να μάθετε αν είναι στη φυλακή, να τα αναφέρετε, να, να ξέρετε περί τίνος πρόκειται, έτσι σε πιο μικρές ομάδες και πολύ τεχνικό ε, τρόπο μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τους εμπειρογνώμονές μας στις Βρυξέλλες για κάθε χώρα. Και τέλος, αν υπάρχει κάποια δράση από την Επιτροπή σας ή από το Κοινοβούλιο που θέλετε να έχετε ομιλητή από κάποια χώρα, μπορούμε επίσης να υποστηρίξουμε. Ιδιαίτερα αν πρόκειται για δικαιούχους που παίρνουν χρήματα από εμά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διαφωτιστική αυτή παρουσίαση που κάνατε και πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό για μας να ακούμε την παρουσίαση αυτή μετά από τις μαρτυρίες που ακούσαμε από δύο υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων σήμερα το πρωί. Νομίζω λοιπόν ότι η δική σας συμβολή θα είναι πραγματικά πολύτυπη. Έχουμε ήδη καθυστερήσει, όμως φταίω εγώ ως νέα προεδρεύουσα εδώ στην Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε πάντως για την ιδιαίτερα αυτή ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Να ζητήσω τώρα από τους βουλευτές να είναι σύντομοι στις παρεμβάσεις τους. Ιζαμπέλ πρώτη, ξενόματος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω, κύριε Πομιανόφσκι, για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση που κάνατε. Νομίζω ότι αν δεν είχε εκπονηθεί το Ταμείο αυτό, αν δεν είχε αναλάβει δράση, θα έπρεπε να το δημιουργήσουμε σίγουρα από την αρχή. Χαίρομαι πάρα πολύ που είπατε ότι υποστηρίζετε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν καμία υποστήριξη από πουθενά και συνεχίζω στα γαλλικά. Συμπληρώνονται κατά αυτόν τον τρόπο τα εφιστάμενα κενά και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε μία παρέμβαση μη πολιτική, αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική στο ανθρωπιστικό πεδίο, στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένως, θα ήθελα ειλικρινά να σε ευχαριστήσω ολόθερμα και να σας ρωτήσω το ακόλουθο. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε τρόπον την να ενισχύσουμε, συγγνώμη, στα αγγλικά μου έρχεται να ενισχύσουμε τη σχέση που έχουμε με εσάς, αν πιστεύετε εσείς ότι μεταξύ μόνο σχέση μπορεί κάπου και κάπως να ενισχυθεί. Σας ευχαριστώ πολύ να απαντάω σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά, κύριε Πρόεδρε. Θα ακούσουμε ακόμα κάποιε ερωτήσει και θα απαντήσετε στην συνεχεία. Ο Ραφαήλ Γκλουξμάν, σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σα. Όντω, νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Καταπιστευματικό Ταμείο για τη Δημοκρατία είναι μια εξαιρετική ιδέα και ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο δημιουργήθηκε σε μια πολύ διάζουσα ιστορική στιγμή. Αρχικά απευθυνόταν στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης και ουσιαστικά αυτό το οποίο έλειπε ήταν ένα τέτοιο εργαλείο στο πλαίσιο της ήπιας διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρεις ερωτήσεις θα ήθελα να θέσω. Πρώτον, πώς μπορούμε εμείς να σας βοηθήσουμε για να αυξήσετε τον προπολογισμό σας γιατί 60 εκατομμύρια ευρώ έχετε δαπανίσει. Αυτό είναι πολύ θετικό και ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Να μπορούμε να αυξήσουμε τον προπολογισμό και κατά αυτόν τον τρόπο να χρηματοδοτήσουμε περισσότερε δράσει, αυτό θα είναι ακόμα καλύτερο. Δεύτερον, πώ μπορούμε να αυξήσουμε τη σφαίρα επιρροή σα, τη σφαίρα δράση σα. Για παράδειγμα, σε χώρε σαν το Σουδάν, που μόλι πέρασε από επανάσταση, Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι δημιουργούν αυτή τη στιγμή διάφορα κινήματα. Εσείς μπορείτε να βοηθήσετε ανθρώπους σε μια χώρα σαν το Σουδάν. Πώς μπορούμε εμείς να σας βοηθήσουμε προκειμένου να παρέμβετε και σε αυτή τη χώρα. Και τρίτη ερώτηση, ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την επόμενη συζήτηση που θα ακολουθήσει που αφορά την Αλγερία. Ποιες δράσεις έχετε να δείτε εσείς στη χώρα αυτή και τι είδους δυνάμεις υποστηρίζετε εσείς σε αυτή τη χώρα μετά την τεράστια αυτή κινητοποίηση που είχαμε στη χώρα αυτή που βρίσκεται ακόμα βέβαια υπό την επιρροή και την επίδραση των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας. Σας ευχαριστούμε πολύ Ραφαέλ, Τζίνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την παρουσίαση αυτή Προσβλέπω στη συμμετοχή μου στο Προεδρείο εξ ονόματος των Πρασίνων, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία. Ω νέο Ευρωβουλευτή, θα ήθελα να γνωρίζω λίγο περισσότερα για τη δράση σα. Θα ήθελα και εγώ να θέσω τρει ερωτήσει. Είπατε ότι θέλετε να συνεργαστείτε με του γείτονε των γειτόνων. Επομένω, κατά αυτόν τον τρόπο επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογή του Ταμείου σα. Από την άλλη, λέτε όμω θέλετε να είστε ένα εργαλείο ιδιαίτερα ευέλικτο. Αυτό δεν θα επηρεάσει το βαθμό αποτελεσματικότητά σα. Επίση, από όσο κατάλαβα, υπάρχουν ορισμένε χώρε οι οποίε δεν συμβάλλουν στο Ταμείο αυτό, όπω η Γαλλία, αν δεν κάνω λάθο. Ορισμένα κράτη-μέλη δεν συνεισφέρουν στον προπολογισμό του Ταμείου, αλλά πάλι είπαν ότι θέλουν να γνωρίζουν ότι θα χρηματοδοτούνται συγκεκριμένοι τομεί και συγκεκριμένε δράσει αυτό πώς επηρεάζει τελικά την αποτελεσματικότητα του δικού σας του Ταμείου και πώς μπορούμε αυτό να το διορθώσουμε. Και κάτι ακόμα. Το Ισραήλ και η Παλαιστίνη είναι μια περιοχή ιδιαίτερα προσφυλή σε μένα. Μόλι επέστρεψα από μια διακομματική αποστολή που έλεγε χώρα κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών και από ό,τι ε, κατάλαβα, έχετε καταφέρει να υποστηρίξετε κάποιε ομάδε τη κοινωνία των πολιτών μετά την τελευταία εντιφάντα που είχαμε στην περιοχή. Διερωτώμε λοιπόν με τα αποτελέσματα επίσης ε, των εκλογών όπως τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή ενδεχομένως τα πράγματα να επιδεινωθούν ακόμα περισσότερο. Η δική σας η προσέγγιση ποια είναι. Θα μπορούσαμε να επέμβουμε και στην ε, περιοχή αυτή για να βελτιώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση μέσω του Ταμείου σας ενώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε σύντομο, σας παρακαλώ πολύ, γιατί πρέπει να δώσουμε και το λόγο τα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ιδιαίτερα θετικές οι ερωτήσεις σας, γιατί ξεκινήσατε όλοι με πολύ ενθαρρυντικά λόγια. Μας είπατε να συνεχίσουμε το έργο μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τα σχόλιά σας αυτά. Για να απαντήσω καταρχάς στην ερώτηση της ε, Ιζαμπέλ. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο περιστασιακή δράση μας, έχει και μια πολιτική φύση. Ξέρετε ότι ακόμα και όταν επεμβαίνουμε για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η επέμβασή μας αυτή έχει μια έντονη πολιτική φύση, μια έντονη πολιτική απόχρωση. Να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπερασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς να επεμβαίνουμε με κάποιο πολιτικό τρόπο τελικά. Τα δύο, οι δύο πτυχές αν θέλετε συνδέονται μεταξύ τους. Γι' αυτό το λόγο και η σχέση που έχουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί εσείς είστε αν θέλετε η πολιτική δύναμη της Ευρώπης. Και δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση μπορούμε να σχετικοποιήσουμε τη σημασία που έχει για την πολιτική η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχω διαβάσει διάφορες δηλώσεις που έχουν κάνει συναδελφοί μας από τις Ηνωμένε Πολιτείε. που αναφέρονται ουσιαστικά στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι τελικά υποστηρίζονται πάρα πολύ, αναβαθμίζονται από τις δηλώσεις που γίνονται ή που μπορούν να γίνουν σε πολιτικό επίπεδο. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή λένε ότι δεν έχουν την απαραίτητη υποστήριξη, ότι ουσιαστικά δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα σε αυτά τα οποία λέμε θεωρητικά και σε αυτά τα οποία κάνουμε στην πράξη. Ελπίζω ότι τουλάχιστον στην Ευρώπη θα φροντίσουμε να συνδυάσουμε περισσότερο τις πολιτικές δηλώσεις με την επιτόπου δράση. Η επιτόπου δράση, η επιτόπου παρέμβαση θα πρέπει να στηρίζεται από τις αντίστοιχες πολιτικές δηλώσεις. Όσον αφορά την μεγαλύτερη συλλογή πόρων, προφανώς μπορείτε να βοηθήσετε. κάθε χώρα που εκπροσωπείτε εδώ πέρα είναι ένας δυνάμει χορηγός του Ταμείου μας. Ξέρετε ότι πολλέ φορέ οι χώρε και οι κυβερνήσει δεν αποφασίζουν από μόνε του για την χρηματοδότηση αυτή. Πολλέ φορέ πρέπει να του ασκηθεί πίεση πρώτα, ακόμα και από του εκλεγμένου όπω είστε εσεί, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν ένα ταμείο το δικό μα. Τώρα, μακρά ιστορία έχουμε με τη Γαλλία. Αρχικά η Γαλλία ε, ήταν πάρα πολύ διστακτική ακόμα και για την ίδια τη θέσπιση του ταμείου αυτού έχει αλλάξει πλέον τη στάση της. Τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια έχουμε έναν πολύ έντονο διάλογο με το Υπουργείο Εξωτερικών στη Γαλλία, με τους αρμοδίους στο Παρίσι. Δεν έχει ληφθεί όμως ακόμα μία απόφαση χρηματοδοτικής συνδρομής ε, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία. Ακόμα περιμένουμε λοιπόν. Θα λέγω ότι εν γέννη τα κράτη-μέλη της Μεσογείου, από την περιοχή της Μεσογείου δεν έχουν δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ στη χρηματοδότηση του Ταμείου με την εξαίρεση της Ισπανίας η οποία χρηματοδοτεί το Ταμείο. Σαφώς λοιπόν μπορούμε να αναλάβουμε δράση για να διορθώσουμε την κατάσταση και βέβαια εσείς οι ευρωβουλευτές μπορείτε να βοηθήσετε ιδίως στις διμερείς επαφές που έχετε με τους αρμοδίους στις χώρες αυτές. Όσον αφορά τώρα το Σουδάν και την Αλγερία, Ξέρω ότι οι περιοχές αυτές και η πολιτική του κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, Επομένω μπορούμε να σας δώσουμε και πιο λεπτομερεί πληροφορίες διμερώς. Γνωριζόμαστε πολύ καλά, επομένω μπορούμε να σας διαβιβάσουμε τις πληροφορίες αυτές. Έχουμε προγραμματική περισσότερο στην Αλγερία και λιγότερα στο Σουδάν και στις δύο χώρες έχουμε μια ευαίσθητη πολιτική κατάσταση οι χώρες αυτές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την πολιτική υποστήριξη και υπάρχει μια ευαισθητοποίηση σε σχέση με αυτό. Υπάρχουν φορείς οι οποίοι μπορεί να στιγματιστούν μόνο και μόνο επειδή δέχονται υποστήριξη απ' έξω, από το εξωτερικό. Πρέπει λοιπόν στην παρέμβασή μας στις χώρες αυτές να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην εκθέσουμε κάποιους εκεί τοπικούς παράγοντες. Ασχολούμεθα πάντως και με τις δύο αυτές ε, χώρες και θα θέλαμε να ενισχύσουμε τον ε, διάλογο που έχουμε και στην περίπτωση της Αλγερίας, όπως σας είπα, ήδη υπάρχουν κάποια προγράμματα σε εξέλιξη, ενώ συζητούμε αυτή τη στιγμή για τη δυνατότητα εφαρμογής κάποιων προγραμμάτων στο Σουδάν. Όσον αφορά τώρα τη χρηματοδότηση εκ των προτέρων συγκεκριμένων προγραμμάτων, συγκεκριμένων δράσεων, αυτό έχει αποτελέσει πρόβλημα θα πρέπει τώρα εμεί στην γραμματεία του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία, από το να έχουμε ένα συλλογικό ταμείο, το οποίο να χρηματοδοτεί γενικά και όριστα προγράμματα, να μπορούμε να έχουμε μια κατάτμιση του προπολογισμού μα και να φαίνεται ξεκάθαρα εξ αρχή ποια γραμμή του προπολογισμού χρηματοδοτεί ποιο πρόγραμμα. Το πρόβλημα είναι ότι ε, είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή στα πλαίσια του Δυτικού Συμβουλίου να κάνουμε μια τέτοια αλλαγή. Συμμετέχοντας κάποιος πάντως στο Λογικό Συμβούλιο μπορεί να θέσει κάποιες προτεραιότητες, αλλά δεν θα θέλαμε αυτή τη στιγμή να περιορίσουμε συγκεκριμένα τμήματα του προπολογισμού για συγκεκριμένες μονοδράσεις και να δεσμεύσουμε κατά αυτόν τον τρόπο εκ των προτέρων συγκεκριμένα τμήματα του προπολογισμού. Πάντως, είναι μια πρόκληση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο επειδή υπάρχει έλλειψη κατανόηση ή ακόμα και πολιτική βούληση, αλλά πολλέ φορέ επειδή και ο ίδιο ο δημοσιονομικό μα κανονισμό ή κανονισμοί, οι δημοσιονομικοί, οι κανονισμοί επί του προπολογισμού συγκεκριμένων κρατών μελών δεν μα επιτρέπει μια τέτοια χρηματοδότηση. Μια χρηματοδότηση γενική δηλαδή, η οποία δεν θα είναι εκ των προτέρων διαιρεμένη σε συγκεκριμένα τμήματα, συγκεκριμένε γραμμέ προπολογισμού και συγκεκριμένε δράσει. Αν καταλήξουμε σε ένα τέτοιο τελικά σύστημα, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να διχειριστούμε διαφορετικά την κατάσταση, να έχουμε εξ αρχή διαφορετικά κονδύλια για διαφορετικά προγράμματα και να έχουμε και μια ομάδα που να ασχολείται με τον, με τον προπολογισμό με αυτή τη μορφή. Όσον αφορά το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, έχουμε προγράμματα και στι δύο περιοχέ. Πρέπει να σα πω ότι ορισμένα από τα προγράμματά μα, για παράδειγμα στο Ισραήλ, κέντρισαν το ενδιαφέρον της προηγούμενης κυβέρνησης, όχι με θετικό θα έλεγα τρόπο, χωρίς όμως και να έχουν αναλάβει κάποια επιθετική στάση απέναντί μας, αλλά ακούσαμε και κάποια επικριτικά σχόλια από κάποιους Ευρωπαίους αξιωματούχους, πολιτικούς μάλλον, ότι ενδεχομένως να υπερβάλλουμε λίγο προσπαθώντας να σκαλίσουμε και να διερευνήσουμε συγκεκριμένες δημοκρατικές αδυναμίες ή κάποια δημοκρατικά ελλείμματα στο Ισραήλ. Πάντως νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό επίπεδο αξιοπιστία απέναντι στην Παλαιστίνη και άλλες αραβικές χώρες. Όταν λοιπόν υπάρχει κάπου ένα δημοκρατικό έλλειμμα, αυτό θα πρέπει εμείς να το τονίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο για ένα δεύτερο γύρο, αν υπάρχουν επιπλέον ερωτήσει. Εάν όχι, θα δώσω το λόγο στην κυρία Γιούλια Ρούπε, που είναι υπεύθυνη για θέματα δημοκρατίας και εκλογικής παρατήρησης ε, και αποστολές εκλογικής παρατήρησης στην ε, υπηρεσία εξωτερική δράση Και εσεί για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ, κύριε ε, Πομινόφσκι, για την παρουσίασή σα. Ε, η υπηρεσία, μα, η υπηρεσία σας συνεχίζει να είναι ένας αξιόπιστος εταίρος με τις ε, διαρκείς, ε, σωστές και ταχύες πληροφορίες που μας παρέχεται. Πολλές φορές τα στοιχεία που μας παρέχεται είναι πολύ σημαντικά για όλους τους δωρητές, Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη-μέλη. Ένας από τους βασικούς τομείς που ε, μπορούμε να προσφέρουμε και μας βοήθεια είναι τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ε, μαζικής ενημέρωσης. Η ραχοκοκαλιά της δημοκρατίας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη λογοδοσία και την προσφορά καλής πληροφόρησης στους πολίτες και τους πολιτικούς ηθήνοντες. Και σε εμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπηρεσία, μας έχει κάνει πολλή δουλειά για να υποστηρίξει τα ε, ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης Μήπως θα μπορούσατε λίγο να επιβραδύνετε για τους διερμηνείς. Με την διερεύνηση ε, στο διαδίκτυο από νέους δημοσιογράφους ή καινούριους δημοσιογράφους, ε, ώστε να παραμένει ανεξάρτητο αυτό το πολυφωνικό πλαίσιο. Προσπαθούμε να πλησιάσουμε τους νέους και την διασπορά τους μετανάστες διαφορών χωρών Θέλουμε να έχουμε μακροπρόθεσμη υποστήριξη και ακριβώς για αυτό το λόγο η υπηρεσία μας δεν μπορεί να γίνει ένας εταίρος ε, διαρκείας για τα περισσότερα μέσα. Αναζητούμε λοιπόν ε, μέσα, ε, πρωτοβουλίες που έχουν υποστηριχθεί με επιτυχία ως τώρα από το καταπίστευμα. Μα ενδιαφέρει επίση τι δωρέ έχουν δοθεί και σε συγκεκριμένε επιχειρήσεις ε, στις ε, χώρες με τι οποίε συνεργαζόμαστε. Με το καταπίστευμα και το Ευρωκοινοβούλιο θέλουμε από την υπηρεσία μας να δούμε πώς μπορεί να ε, εξεταστεί το θέμα της διαρκούς υποστήριξης. Θέλουμε επίσης να συνεχίσουμε την συνεργασία μας με, την, με το καταπίστευμα και με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα αναλάβει σύντομα, τη Νέα Προεδρία εννέα βουλευτές πρόκειται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μας ενδιαφέρει πολύ να δούμε τι επιλογή θα γίνει ώστε να ασχοληθούμε όλοι μαζί για τα, με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία. Ελπίζουμε να συμμετέχουν και μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστούμε. Οπότε εδώ να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Κύριε Πομιονόφσκη, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα διαφωτιστική η παρουσίασή σας και νομίζω ότι όλη σας προσέγγιση τουλάχιστον για μένα ήταν ιδιαίτερα λογική. Σημείωσε και τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να σας βοηθήσουμε να είστε βέβαιος ότι μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μας. Ευχαριστώ.